σήμερα το πρωί ότι δεν θεωρεί ότι το θέμα πρέπει να τεθεί στη σημερινή ημερήσια διάταξη. Και αυτό έπρεπε να σας το ανακοινώσω. Ο κύριος Λάμπερτς έχει το λόγο. Ευχαριστώ για τις εξηγήσεις σας, Πρόεδρε. Ε, προφανώς υπάρχουν πολλοί που δεν επιθυμούν να συζητηθεί η κατάσταση στη Δανία. Πιστεύω όμως ότι πρόκειται για, το, για θέμα αξιοπιστίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και γι' αυτό το λόγο η, ε, η συνθήκη ε, απαιτεί να είμαστε δίκαιοι. Ε, χτες ε, αφιερώσαμε ένα σημαντικό χρονικό διάστημα στην κατάσταση στην Πολωνία και πολύ σωστά. Ήταν σωστό και δίκαιο. Το ίδιο και με την Ουγγαρία. Αυτή τη στιγμή έχουμε μια κατάσταση εν εξελίξη στη Δανία που απαιτεί να τη συζητήσουμε, κατά την άποψή μου. Στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών ε, ε, θα έπρεπε να συζητηθεί το θέμα αυτό πριν τη συζήτηση στην Ολομέλεια. Όμως, ε, τα μέλη της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών αρνήθηκαν να συζητήσουν εγκαίρως τα μέτρα αυτά πριν εγκριθούν από το Κοινοβούλιο της Δανίας. Γι' αυτό το λόγο σας ζήτησα το θέμα να συζητηθεί στην ε, Ολομέλεια. Εσείς λέτε ότι μιλήσατε με τους εκπροσώπους των πολιτικών ομάδων, αλλά εγώ σας ζητώ το θέμα να ψηφιστεί από εμάς εδώ στην Ολομέλεια, γιατί γνωρίζω ότι στο εσωτερικό των πολιτικών ομάδων υπάρχουν πολλοί που θέλουν το ζήτημα αυτό να συζητηθεί στην Ολομέλεια ε, ε, κατά τη διάρκεια αυτής της συνεδρίας. Οπότε ζητώ να θέσετε το θέμα σε ονομαστική ψηφοφορία εδώ και τώρα. Για να δούμε αν χάνουμε ή κερδίζουμε. Η κυρία Τσίμα. Κύριε Πρόεδρε, υποστηρίζω το αίτημα του κύριου Λάμπερτς και πρέπει να πω πως έχω ενοχληθεί και απορώ η διάσκεψη των Προέδρων όσον αφορά το αίτημα των Πρασίνων που ετέθη για να ασχοληθούμε με το θέμα αυτή την ε, εβδομάδα το υπό την αίρεση το ότι θα συνεδρίαζε η Επιτροπή Λίμπε την Δευτέρα που μας πέρασε τελικά το απέριψε αλλά τελικά νομίζω πως ήταν σαφές ότι θα το συζητούσαμε ούτως ή άλλος ανεξαρτήτως του τι θα κάναν οι συντονιστές ή η Επιτροπή ΛΥΜΠΕ. Θα ήθελα λοιπόν και εγώ να γίνει μια ε, ψηφοφορία. και νομίζω πως ε, υπάρχει η δυνατότητα να το συζητήσουμε αυτή την ε, στιγμή. Εκτό αν ο μόνος σα στόχο είναι να μην ε, το συζητήσουμε εδώ πέρα πριν ληφθεί οποιαδήποτε απόφαση στο Κοινοβούλιο της Δανία. Σας ευχαριστώ κυρία Ίνετφελτ. Σας ευχαριστώ. Η ομάδα μου συμφωνεί ότι είναι σημαντικό να συζητηθεί αυτό το θέμα σε αντίθεση με τα όσα νομίζει ο κύριος Λάμπερς και η κυβέρνηση της Δανίας θέλει να έρθει εδώ πέρα να το συζητήσει το θέμα. Ήταν διατεθειμένοι να έρθουν και αυτή την εβδομάδα. Ναι, είναι σημαντικό να το συζητήσουμε πριν ψηφιστεί στο Κοινοβούλιο της Δανίας, αλλά είναι κάπως τεχνητό τώρα να πιέζουμε για μια συζήτηση αυτή την εβδομάδα σε αυτή την ολομιλία. Αλλά υπάρχει η δυνατότητα, την Δευτέρα υπάρχει άλλη συνεδρίαση της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ και θα ήθελα να σας παρακαλέσω κύριε Πρόεδρε να έρθετε ξανά σε επαφή με τον Πρόεδρο και τους συντονιστές της Επιτροπής Ελευθεριών και να τους ε, ζητήσετε να το βάλουν στην ημερήσια διαταξή της Δευτέρας. Ευχαριστώ. Ο κύριος Βέμπερ. Κύριε Πρόεδρε, ήδη τη Δευτέρα όταν παρουσιάσατε την ημερήσια διάταξη αυτή τη εβδομάδα, σα ανέφερα τη θέση του ΕΛΚ. Και τώρα ισχύει το εξή. Εδώ υπάρχουν οι πυρογνώμονε, οι συνάδελφοι από την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, οι συντονιστέ, όλοι αυτοί που έχουν οριστεί αρμόδιοι για θέματα εσωτερικών υποθέσεων. Αυτοί λοιπόν διαβουλεύτηκαν και αποφάντηκαν ότι το θέμα δεν είναι επίγον. Και θεωρώ ότι οι πράσινοι θα πρέπει να σεβαστούν το ότι οι εμπειρογνώμονε του Κοινοβουλίου ότι το θέμα δεν είναι επίγον. Η κυβέρνηση της Δανίας με ε, κατηγορηματικότητα ανέφερε ότι είναι πρόθυμη να έρθει εδώ να συζητήσει. Γι' αυτό λοιπόν ε, θα πρέπει να αφήσουμε τους συναδέλφους μας ε, να δουλέψουν κανονικά. Και θέλω σήμερα να πω το εξής. Όσον αφορά την νομοθεσία ή την πρόταση στη Δανία, είναι το θέμα το εξή. Ε, οι ε, ε ζητούντες, ε, άσυλο είναι εξισώνονται με τους δανούς γιατί υπάρχουν και δανείοι που είναι φτωχοί και δεν έχουν χρήματα. Στο μέλλον λοιπόν κύριε Λάμπερτ, αν οποιαδήποτε νομίζετε επιτάπητος θέλουμε αυτούς που την θέτουν να τους επισημάνουμε ποια είναι η ιδεολογία των πρασίνων αν το κάνουμε αυτό στο μέλλον τότε θα ζημιώσουμε το ευρωπαϊκό εγχείρημα. Η δική μου πολιτική ομάδα σέβεται όλα αυτά αυτά που ε, λαμβάνουν χώρα στο Κοινοβούλιο της Δανίας. Έχει ζητήσει το λόγο ο κύριος Βιστίζεν, ο κύριος Γκερέρος Σαλόμ και νομίζω ότι μετά πρέπει να ληφθεί μια απόφαση. Ο κύριος Βιστίζεν έχει το λόγο. Θα ήταν παράλογη επίδειξη ισχύω από πλευράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αν ξεκινούσαμε να παρεμβαίνουμε στις εργασίες του Δανεισικού Κοινοβουλίου. Ε, εμείς ε, έχουμε επιβεβαιωθεί από τους ψηφοφόρους. Σε κάθε περίπτωση η Δανία είναι μια δημοκρατία και μόνο η Κομισιόν και ο κύριος Τίμερμανς και όχι η ομάδα των Πρασίων στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που θα έπρεπε να ερευνήσουν τα όσα κάνει η κυβέρνηση της Δανίας. Τρίτον, πρόκειται για ένα νομοσχέδιο. Δεν έχει υιοθετηθεί ακόμα από το Κοινοβούλιο της Δανίας. Από την πρώτη ανάγνωση βέβαια γνωρίζουμε ότι έχει γίνει πολύ θετικά αποδεκτό. Ε, υποβλήθηκε από το ε, κόμμα της Δανίας και ε, έχει υποστηριχθεί και από το Λαϊκό Κόμμα και από άλλα κόμματα του Κοινοβουλίου. Οπότε δεν θα πρέπει να παρέμβουμε ε, στα εσωτερικά της Δανίας. Ε, Ο κ. Γκερέρο. Ε, η ομάδα μου προτιμά να στηρίξουμε την πρόταση του, ε, της διάσκεψης των Προέδρων και την απόφαση της πλειοψηφίας της Επιτροπής ΛΥΜΠΕ. Παρ' όλα αυτά δεν συμφωνώ απόλυτα με όλα τα επιχειρήματα τα οποία ε, προβλήθηκαν ε, τώρα, πριν από λίγο. Πιστεύω ότι η κατάσταση στη Δανία αξίζει να συζητηθεί σε βάθος από το Ευρωπαϊκό Κοινοβουλίο και ακριβώς για αυτό το λόγο, ακριβώς για αυτό το λόγο πιστεύω ότι δεν θα πρέπει να γίνει με αυθόρμητο και ανοργάνωτο τρόπο. Θα πρέπει να γίνει μια συζήτηση στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών καταρχήν και αργότερα στο, στην Ολομέλεια οργανωμένα. Vielen Dank, Ευχαριστούμε πολύ κύριε Γκερέρο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, νομίζω ότι είναι σαφής η εικόνα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Υπάρχει σαφήνεια. Ο κύριος Λάμπερτς ε, θέλει να ψηφίσουμε για το κατά πόσον θα πρέπει να συζητηθεί το θέμα στην Ολομέλεια σήμερα ή αύριο. Η κυρία Ινφελτ προτείνει η κυρια προτείνει προτεινει επιτροπη Ελευθεριών να συζητήσει το θέμα τη Δευτέρα, την επόμενη Δευτέρα. Αυτές είναι δύο διαφορετικές προτάσεις που έχουν κατατεθεί και νομίζω ότι η πλειοψηφία τάσεται υπέρ της πρότασης της κυρίας Ιντφελτ. Νομίζω είναι σαφές αυτό. Ξέρω κύριε Λάμπερτς ότι διαφωνείτε, το έχω καταλάβει, το έχω καταλάβει απόλυτα. Αλλά ξέρετε η δουλειά του Προέδρου είναι να ε, βολιδοσκοπεί ποιε είναι οι διαμορφούμενε ε, πλειοψηφίε. Λοιπόν, πρώτα να ψηφίσουμε για την πρόταση τη κυρία Ιντφελτ. Αλλά πριν έχει δει το λόγο ο κύριος επί διαδικαστικού. Ευχαριστώ. Ο κανονισμό βασίζεται στα άρθρα 150 και 154 για τη συγκεκριμένη περίπτωση. Σε κάθε περίπτωση δεν είναι δυνατόν δεν θα ήταν δυνατόν να τεθεί σε ψηφόρια οποιαδήποτε πρόταση. Το άρθρο 152 είναι σαφές. Ε, λέει ότι η μέση διάταξη της ε, Συνόδου υιοθετείται στην αρχή της Συνόδου. Υπάρχει δυνατότητα βέβαια εκ των υστέρων τροποποίησης με επιβάση του άρθρου 154 για περίπτωση επίγοντο θέματος. Όμως αυτή θα πρέπει να ε, παρουσιαστεί από τον πρόεδρο να μεταφραστεί σε όλες τις γλώσσες και είναι δυνατόν να συζητηθεί μόνον στην επόμενη σύνοδο που αυτήν παρουσιάζει το σημείωμά του Πρόεδρος. Συνεπώς η διαδικασία η οποία έχει ακολουθηθεί ε, θα ήταν έτσι κι αλλιώς ε, σε αντίφαση με τον κανονισμό μας ε, αν ψηφορία το θέμα βέβαια. Κύριε Γκολνίς, ε, από ό,τι φαίνεται διαβάζετε το κανονισμό του Κοινοβουλίου, αλλά δεν, καταλαβαίνετε, δεν το καταλαβαίνετε καλά, δεν τον ερμηνεύετε σωστά. Ο πρόεδρος μπορεί να προτείνει να αλλάξει η ημερήσια διάταξη. Αυτή η προνομία υπάρχει για τον πρόεδρο του Κοινοβουλίου. Μπορώ δηλαδή, έχω το δικαίωμα να προτείνω και γι' αυτόν ακριβώ το λόγο εχθέ το βράδυ παρακάλεσε τι πολιτικέ ομάδε να μου ανακοινώσουν ποια είναι η άποψη των πολιτικών ομάδων επί του θέματο. Και η διαβούλευση κατέληξε σε μια αδιαμφισβήτητη πλειοψηφία. Η πλειοψηφία λοιπόν τάσεται υπέρ του να μην αλλάξει η ημερήσια διάταξη. Και γι' αυτό δεν είχα προτείνει αλλαγή. Τώρα, είναι άλλο θέμα το κατά πόσον ένα μέλο του Κοινοβουλίου που ε, υποβάλλει την πρόταση η Ολομέλεια να συστήσει να επιληφθεί μια επιτροπή του θέματος. Αυτή είναι η πρόταση της κυρίας Ιντφελτ που δεν έχω κανένα πρόβλημα να την παρουσιάσω και γι' αυτό λοιπόν σας είπα και προηγουμένως προτείνω να ψηφίσουμε επί της πρότασης της κυρίας Ιντφελ. Ο κύριος Λάμπερτς. Δεδομένου ότι ήταν πρόταση ε, της ε, διάσκεψης των Προέδρων, θα ήθελα αυτή αυτήν την πρόταση να θέσουμε σε ψηφοφορία. Δηλαδή, ε, έτσι κι αλλιώ, ε, εμεί το ζητήσαμε πρώτοι. Ε, να θέσετε σε ψηφοφορία τη δική μα πρόταση και αν απορριφθεί, να τεθεί σε ψηφοφορία η πρώτη κυρία Σίντβελτ. Κύριε Λάμπερτ, αντιλαμβάνομαι την θέση σα, αλλά έχω διαφορετική άποψη. Αν υπάρχει αίτημα στην Ολομέλεια ότι θα πριν συζητηθεί κάτι στην Ολομέλεια να πάει ε, σε μια επιτροπή πρέπει να το ε, ψηφίσουμε. Αν λοιπόν η πλειοψηφία είναι να το συζητήσουμε εδώ πέρα, ναι βεβαίως. Να ψηφιστεί. Λοιπόν, το αίτημα είναι το εξής. Να, ζητήσουμε, να ζητηθεί από την ε, Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών να συζητήσει το θέμα τη δεύτερη μας έρχεται. Ποιος είναι υπέρ. Κατά. Αποχές. Ηλεκτρονική ψηφοφορία. Υπέρ του αιτήματος Ινετφέλτ. Για την, πολιτική, για την Επιτροπή Ελευθεριών. Λοιπόν, πέρας. Γίνεται δεκτό λοιπόν το αίτημα. Σας ευχαριστώ. Περνάμε τώρα. Στο πρόγραμμα δραστηριοτήτων της Ολλανδικής Προεδρίας ο Προεδρεύων ε, έχει τον λόγο, ο Πρωθυπουργός του Βασιλείου των Καταχωρών. Κύριε Μάρκο Ρίτο, έχετε τον λόγο. mr